Θα πρέπει γρήγορα να εθετηθεί το μέτρο και θα πρέπει να κάνουμε το δυνατόν να περάσει το μέτρο το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε αύριο, λέει ο Πρόεδρος, στις 12. Πάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης την έκθεση Κιστόλτ Ρόβολτ όσον αφορά την αυτόνομη δασμολογική ποσόστοση για τις εισαγωγές βοηού κρέατος υψηλής ποιότητας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κριστόλτ Ρόλ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συναδελφοί. Μια εμπορική διαμάχη 14 ετών αύριο θα λάβει τέλος με την ψηφοφορία αυτής της έκθεσης. Η διαφωνία αυτή οφείλεται σε μία απόφαση του 1998 του ΠΟΕ καθώς έκτοτε αναγκαστήκαμε, τον όπως του λέγει, να εισάγουμε κρέας ε, με ορμόνες από τις ΙΠΑ. Τέλος πάντων, ε, δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν και για τις κυρώσεις, απλά θέλω να πω πως χαίρομαι για το ότι καταφέραμε να τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση. Η Προεδρία της Δανίας, εξ ονόματος του Συμβουλίου, ήδη έχει συμφωνήσει σε άτυπο τριμερή διάλογο με την έκθεσή μου, οπότε δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο και να τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση. Οπότε θα ήθελα με βάση τα όσα σας είπα να συμφωνήσετε και να υπερψήσετε ναι είναι ένα συμβιβασμό, αλλά ο συμβιβασμό αυτός κατά, ε, κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ ισορροπημένος. Και ιδιαίτερα τώρα η ευρωπαϊκή ε, γεωργία θα μπορεί να προγραμματίζει καλύτερα κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο. Επιπλέον, πέρα από αυτή την έκθεση υπάρχει εδώ πέρα ένα σημάδι, ένα μήνυμα για τις υπερατλαντικές σχέσεις. Έχουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιες διαφορές απόψεων και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε από κοινού διεθνή πρότυπα. Δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Μόνο η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού θα μπορέσουν να σταθούν στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του αύριο. Οπότε καλωσορίζω επίσης το ότι για παράδειγμα τώρα έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τις δουλειές και την ανάπτυξη όπου θέλουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε η ανάπτυξη πράγματι να ε, υπάρξει. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο όσον αφορά το μέλλον. Από τις ε, εποχές της ε, σπογκώδους εγκεφαλοπάθειας η ΕΠΑ επέβαλαν απαγόρευση εισαγωγής βοήου κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο όμως δεν θεμελιώνεται επιστημονικά, καθώς εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις ε, σπογκώδους εγκεφαλοπάθειας ε, των βοηδών. Πρόκειται καθαρά για προστατευτισμό από πλευράς ΙΠΑ. Κυρίες μου και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό στη διάρκεια αυτής της ε, νομοθετικής διαδικασίας ε, πήθηνα επιστολές ε, σε όλους τους ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους και είχα και κάποιες συνομιλίες ειδικά με τον Υπουργό Γεωργίας Βουλσακ και τον Κέρκ, τον εκπρόσωπο του εμπορίου, τους, από τους οποίους ζήτησαν να σταματήσουν αμέσως αυτές οι απαγορεύσεις εισαγωγών και μπορώ να σα ανακοινώσω ένα ευχάριστο νέο, το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. 9 Μαρτίου, την Παρασκευή που μας πέρασε, το Υπουργείο Γεωργίας, τον είπα, δημοσίευσε το λεγόμενο draft call στην ε, υποχρεωτική ε, διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για να αρθεί ε, η απαγόρευση εισαγωγή, ε, καθώ πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα. Οπότε θα ήθελα να σα παρακαλέσω να μην διακινδυνεύσουμε τώρα αυτό το κλίμα συνεργασία το οποίο υπάρχει. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς. Να ευχαριστήσω εδώ πέρα και την Κομισιόν και την Προεδρία του Συμβουλίου για την καλή συνεργασία. Αλλά κυρίως... Ναι, ναι, ναι κύριε Πρόεδρε, είναι 30 δευτερόλεπτα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργίας. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας, γιατί δεν ήταν όλα τα βήματα αυτής της διαδικασίας απλά. Αλλά ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Σιόλος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως την εισηγήτρια, όλα τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για την εργασία τους και την δέσμευσή τους να καταλήξουμε στη συμφωνία, όπως ανέφερε και η εισηγητρία. Η πρόταση αύξησης των δεσμολογικών ποσοστώσεων βοήου χωρίς ορμόνες προβλέπεται από το Μνημόνιο εργασία το οποίο υπογράψαμε με τις ΗΠΑ το 2009 και με τον Καναδά το 2011. Το Μνημόνιο αυτό συνεργασία προβλέπει την προσφορά αμοιβαίω ευκαιριών εκατέρωθεν του Ατλαντικού και αυτό είναι και μια σημαντική εξέλιξη για να θέσουμε τέλος σε μια διαφορά που σοβεί επί δεκαετίες. Οι ΗΠΑ πάβουν τις κυρώσεις κατά ευρωπαϊκών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σημαντική αύξηση της πρόσβασης των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά βοηού κρέατος, χωρίς ορμόνες. Η εισηγήτρια και η αρμόδια επιτροπή υποστηρίζουν την συμφωνία. Η φάση υπορθμών 2 θα δρομολογηθεί τον Αύγουστο του 2012 και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό λύνουμε Οριστικό και μετακλήτω την διαφορά αυτή που είχε πάει και στον ΠΟΕ. Έχω επίγνωση του γεγονότο ότι οι εξαγωγέ βοήου εκατέρωθεν μπλοκαρώνται λόγω των αμερικανικών περιορισμών με πρόσχημα, όπως είπε και η συγγήτρια, την σπογγονδή εγκεφαλοπάθεια των βοηδών. Ο περιορισμός αυτό δεν συνάδει με τη στάση του Διεθνού Οργανισμού Επιζωτιών που πρεσβεύει ότι πρέπει οι εξαγωγέ αυτέ να επιτρέπονται όταν πρόκειται για τι ίδιε κατηγορίε κινδύνου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται ακριβώ στην ίδια κατηγορία κινδύνων που είναι οι ελεγχόμενοι κίνδυνοι. Πρόσφατα συναντήθηκα με τον αναπληρωτή του κ. για να προχωρήσουμε στον, στην αμοιβαία γνώριση των κανόνων βιολογικής γεωργίας. Εκατέρωθαν και ζήτησε από τους Αμερικανούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να σημειωθεί πρόοδος και στον τομέα του περιορισμού των εισαγών βοηού κράτους από την Ευρώπη. Το σχέδιο κανόνων επί του θέματος γνωρίζω ότι ήδη δημοσιεύθηκε το Federal Register στις 9 Μαρτίου. Πρόκειται για δημοσίευση η οποία δρομολογεί διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο μέρος και συνεπώς ανοίγει ο δρόμος, όπως είπε, για τη διευκρίνηση αυτού του θέματος που θα έπρεπε να διευκρινιστεί, όπως προείπε, με βάση τις διεθνές προδιαγραφές. Και επί αυτού του θέματος, λοιπόν, θα καταλήξουμε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα η παραγωγή βοήου εκατέρθεν του Ατλαντικού να μπορούν να απολαύουν αυξημένης πρόσβασης και στις δύο αγορές. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ την Επιτροπή Ίντα και ευχαριστώ και την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων καθώς και το Κοινοβούλιο εν γέννη για την αμέριστη και αποτελεσματική υποστήριξη αυτού του σχεδίου κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε για την Επιτροπή Γεωργίας. Για ένα μισή λεπτό, ο κύριος Λάιον. Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, όπως ο συνάδελφος ο συγγητής από την Ίντερ ανέφερε, 14 χρόνια γίνεται εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση βοήου κρέατος που έχουν υποστεί επεξεργασία μορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσαμε στον ΠΟΕ δύο φορές και υπευλήθησαν και κυρώσεις για τις εξαγωγές από Ευρώπη προς τη ΣΥΠΑ. Αυτό ήταν επιζήμιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη ΣΥΠΑ. Αυτή η συμφωνία που δημοτεύτηκε κάθε άστον το 2009 επιτέλους για μια και καλή άπαξε παντός θα οδηγήσει κάποια λύση. Και νομίζω ότι είναι επικερδές και για τις δύο πλευρές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρείται η απαγόρευση κρεάτων με ορμόνες, βοηού κρέατος με ορμόνες και καταργούνται και οι κυρώσει που είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί στι δικέ μα εξαγωγέ. Σε αντάλλαγμα, η ΕΠΑ έχει 45.000 τόνου πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για βόλιο κρέα υψηλή ποιότητα. Αυτό είναι σημαντικό βήμα πρόοδου. Και εξομάλυνση των σχέσεων των εμπορικών με τη ΣΥΠΑ είναι κάτι πολύ καλό. Ήδη ε, γίνεται κάτι υποφελέ. Σωστά το ανέφερε ο Επίτροπο. Την Παρασκευή ανακοίνωσαν, ΕΠΑ νέου κανόνε τη πογκώδη εγκεφαλοπάθεια για εισαγωγή βοήου. Και ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι απόψε να παροτρύνουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να υιοθετήσει τους νέους κανόνες ε, το ταχύτερο δυνατόν και να αυξηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπορικά θέματα. Αυτό θα είναι επωφελές και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς και για τις Ηνωμένε Πολιτείες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Λάιον. Πάμε στις πολιτικές ομάδες. Για το ΕΛ για δύο λεπτά η κυρία Κέστιγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Θεωρώ πως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή δείχνει πως με αυτή την έκθεση σε αυτό το ακαθόδες θέμα έχει επιτύχει μια, ένα καλό συμβασμό και τη συγχαίρω. Παραμερίζοντας λοιπόν αυτή την διαμάχη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΕ κάνουν ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα. παραμερίζεται έτσι μια εμπορική διαφωνία η οποία είχε ιδιαίτερα αρνητικές ε, συνέπειες μετά από πάρα πολλές ε, αποφάσεις του ΠΟΕ και αμοιβές ε, αμοιβαία εμπορικά αντίπεινα είχαμε οδηγηθεί σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση ενώ τώρα επιτέλους υπάρχει ασφάλεια για τον Ευρωπαίο καταναλωτή αλλά και για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς και η Επιτροπή Γεωργίας στην γνωμοδότησή της ε, είναι ξεκάθαρα υπέρ της υπερψήφισης αυτής της έκθεσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν κρέας με ορμόνες και οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς δεν θέλουν να έχουν εμπόδια στις εξαγωγές τους. Με αυτή λοιπόν την έκθεση έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αμοιβαία υποφελής. Τώρα όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ανοιχτά προβλήματα. Εξακολουθεί να υφίσταται απαγόρευση εισαγωγή του ευρωπαϊκού βοήου κρέατος στη ΣΥΠΑ, το οποίο είναι απαράδεκτο και πρέπει εδώ πέρα να συνεισφέρουμε επικοδομητικά. Θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι να παραμερίζονται οι εμπορικές διαμάχες με τις ε, ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ πέρα μεγάλες ε, προκλήσεις. Πρέπει να φροντίσουμε την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Οι εμπορικέ διαμάχε δεν προωθούν βεβαίως αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς ε, ε, αυτό το οποίο γίνεται είναι πω τελικά τρίτε χώρε καταλήγουν να έχουν καλύτερη θέση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά την εισηγήτρια για την ε, επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Για ένα λεπτό ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ψηφοφορία για το άνοιγμα των δοσμολογικών δασμολογικών ε, ποσοστώσεων για τι αγωγέ βοήου κρέατο υψηλή ποιότητα. Σημαντική στιγμή για την καλή ε, διατλαντική συνεργασία. Για πρώτη φορά, χάρη συνθήκη Λισαβόνα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδες, φορέ την έγκριση τη αποφάσεω αυτή. και θα πρέπει να κατανοήσουν και τα Ηνωμένε Πολιτείε τα θεσμικά όργανα μα. Το είδαμε ότι συναντηθήκαμε στο Κογκρέσο. Μια αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Γεωργία πήγε στι ΗΠΑ. Αυτή η συμφωνία θέτει τέρμα σε μια μακρά και επιζήμια διαμάχη, επιτρέποντα την άρση των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ ε, διατηρώντας ταυτόχρονα την απαγόρευση όσον αφορά τις αγωγές κρέατος με ορμόνες ε, και έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε τα υψηλά επίπεδα προστασία επιστημιστική ασφάλεια και ποιότητα. Γι' αυτό η Επιτροπή Γεωργία που έχω την τιμή να προεδρεύω συμφώνησε απόλυτα χωρί να υπάρξει καμία τροπολογία στην σύναψη αυτή τη συμφωνία, στο πνεύμα της εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων των δύο του Ατλαντικού και να επιλύονται οι διαφορές στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον εισηγητή μας τον κύριο Λάιον. Ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες. 1,5 λεπτό. Η κυρία Σάκη έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κύριε Επίτροπε, από τη συνάδελφη, καλωσορίζουμε την υιοθέτηση αυτή τη έκθεση και θεωρούμε πω τώρα θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα πράγματα. Καθώ αυξάνεται η οικονομική δύναμη των χωρών BRIC, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ΕΕ έχουν αμοιβαίο συμφέρον για να σέβονται του κανόνε του ΠΟΕ. Οι μακροχρόνιες συγκρούσεις όπως αυτή εδώ πέρα η οποία κράτησε σχεδόν 15 χρόνια κάνουν τεράστια ζημιά στις πολυμερείς μα σχέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την απόφαση ως μια αφετηρία για να διευρύνουμε τι σχέσει μας με τις ΗΠΑ και να ζητήσουμε ως κίνηση καλής θέληση από ΣΥΠΑ να άρουν την απαγόρευση για το ευρωπαϊκό βόλιο κρέας. Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη την παγκόσμια διάσταση και κάνοντας αυτό θα πρέπει βεβαίως να μειώσουμε τα εμπορικά εμπόδια και να έχουμε μια διατλαντική αγορά για να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να ξεκινήσουμε στην επόμενη διάσκεψη με τις ΕΠΑ διαπραγματεύσεις για ενιαίο εμπορικό χώρο. Θα πρέπει λοιπόν να βασιζόμαστε σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα και συμπληρωματικότητα. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει όλοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και η Κομισιόν και η Υπηρεσία εξωτερική δράση να προσπαθήσουμε να τους απαθαρρύνουμε από οποιαδήποτε δυσανάλογα μέτρα προστατευτισμού. Οι παρατηρήσεις ε, του Πρόεδρου Σαρκοζή που θέλει να λάβουμε ανάλογα ευρωπαϊκά μέτρα μας δείχνουν τον δρόμο στον οποίο οδηγούμαστε και θα πρέπει να αποφευχθεί. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον στόχο μας και τον ανταγωνισμό για εμπόριο, ταλέντο και αξίες τελικά και θα πρέπει να συνεργαζόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ. μη ένα μισή λεπτό, η κυρία Τόντς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, επίτροπε. Στην Βόρεια Ιρλανδία, στην εκλογική μου περιφέρεια, εξάγουμε γεωργικά προϊόντα. Εξάγουμε περίπου 70% αυτών που παράγουμε και ακόμη περισσότερο στον τομέα του βοηού κρέατος. Συνεπώς, η κυβέρνησή μου αναζητά διαρκώς νέες αγορές αν τα πρόσβαση για το βόλιο κρέας τη Βορειοϊρλανδία. Πρόκειται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία για ένα βήμα προ την σωστή κατεύθυνση. Διορθώνει την αδικία που έγινε κατά των ευρωπαϊκών προϊόντων. Και ελπίζω ότι αυτό θα ισοδυναμεί και με αναγνώριση του υγιεινού φαγητού που παράγουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και το οποίο είναι γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως και άλλοι βουλευτέ προσβλέπω στην σύντομη επίλυση του ζητήματο τη απαγόρευση των ευρωπαϊκών εξαγών λόγω υποτίθεται σπονγκόντου συγκεφαλαιοπάθεια των βοηδών. Ελπίζω ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει στο άνοιγμα και άλλων επιπλέον αγορών για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και δι για το βόλιο κρέας. Κλείνω με μια προειδοποίηση που αφορά τον τομέα του βοήου στην Βορειορλανδία. Οι νέες προτάσεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ συνεπάγονται επιδείνωση για την Βορειορλανδία και το Βόιο οδηγούν σε εντατικοποίηση και επιδείνωση των συνδικών για τους μικρούς παραγωγούς. Ευχαριστώ λίγο Ο λόγος για δύο λεπτά στην κυρία Λεμπρά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πρόκειται για σημαντική συμφωνία η οποία κλείνει αυτές τις μέρες με την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού για την αυτόνομη ποσόστοση για την εισαγωγή κρέατος υψηλής ποιότητας χωρίς Φτάνω λοιπόν στο τέλος μιας εμπορικής διένεξης μεταξύ Ευρώπης αφενός, ε, Αμερικής και Καναδά αφετέρου. Όπως και οι προηγούμενοι μιλητές, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την συναδελφό μου για την σκληρή εργασία τους. Όμως, να ενώσουμε όλοι μας τις φωνές μας για να ταχθούμε υπέρ της υλοποίησης της δεύτερης φάσης. Πρόκειται για νίκη της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Κερδίζουμε τον σεβασμό που αξίζουμε και κατορθώνουμε να επιβάλλουμε οριστικά την απαγόρευση του κρέατος με ορμόνες. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να μας αλλάξουν γνώμη. η απαγόρευση των ευρωπαϊκών εξαγωγών βεβαίω έθεσε σε δινή θέση πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα. Δεδομένου ότι οι δασμοί έφταναν, θυμηθείτε, έως και 300%. Κάτι που ήταν ε, φυσικά ε, αδύνατον να πληρώσουν η παραγωγή του ροκφόρ, των φρέσκων κρεμμυδιών κλπ. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μου τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα βελτιώσει το εμπορικό τη ισοζύγιο και αυτό αποτελεί οξυγόνο για του παραγωγού μα. Εδώ και ένα χρόνο οι Αμερικανοί είδαν όλους τους περιορισμούς, όπως προβλέπετε, οκτώ μήνε δηλαδή πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ήρθε πλέον η στιγμή να πάμε παρακάτω. Οι διαβουλεύσει ήταν επικοδομητικέ, έφεραν αποτελέσματα, απέδειξαν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και καλό όλου να συνεργαστούν δείχνοντας την στάση τους, την διπλωματία τους, τις γνώσεις τους επί τη βάση της αμοιβαιότητας. Αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα δεν αποκλείει το άνοιγμα από το οποίο θα υποφεληθούν και οι δύο πλευρές στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας επιτυχίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Λιμπρά. Δύο λεπτά κυρία Ανδρές. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι πρώτη φορά βάσει τη συνδίκη της Λισαβόνας που το Κοινοβούλιο συμμετέχει σε μια τέτοια συζήτηση με το Συμβούλιο για την έγκριση τροποίησης κανονισμού προϊόν συμβασμού που σχεδιάσαμε πιστεύω πολύ ικανοποιητικά. Καταφέραμε να θέσουμε τέλος σε μια μακροχρονία διαμάχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαγόρευε τη εισαγωγή κρέατο με ορμόνε από τι ΗΠΑ και τον Καναδά. Και οι δύο αυτέ χώρε είχαν επιβάλει εξαιρετικά υψηλού δασμού τη σοκολάτα, το ψωμί, το χείριο κρέα και διάφορα άλλα προϊόντα που έφυγαν τη χώρα μου. Η εξέλιξη λοιπόν είναι ευπρόσδεκτη για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Εμείς διατηρούμε την απαγόρευση εισαγών βοήου με ορμόνες. Από την άλλη πλευρά αυξάνουμε κατά τις εισαγωγές, εισαγω, βοήου κρέατος υψηλής ποιότητας. Στην Ισπανία είχαμε αυτό το 1 εκατομμύριο ε, δασμών. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να εξάγουμε πολύ περισσότερο προ τι ΗΠΑ. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι αντισταθμιστικοί δασμοί που είχαν επιβαλεί οι ΗΠΑ ήταν πάρα πολύ υψηλοί. Τώρα όμω ε, η κατάσταση αυτή τελείωσε. Ήταν υπέρ του Ευρωπαίου καταναλωτή και βεβαίω οδηγεί και σε εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων με τι ΗΠΑ και τον Καναδά. Ένα καλό παράδειγμα, θα έλεγα ένα καλό προηγούμενο για την επίλυση και άλλων παρομοίων προβλημάτων. Ας συνεχίσουμε να επιζητούμε τέτοιου είδου λύσεις σε αντίστοιχα προβλήματα. Ευχαριστώ. Μαγκίνες δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους πολύπους συναδέλφους που εργάστηκαν από αυτού. Ε, όλοι έχουν πολύ καλή διάθεση απόψε γιατί λύσαμε, ελπίζουμε, έναν εμπορικό πόλεμο ο οποίος έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό, 15 χρόνια. Οπότε είμαστε γνώμονες που έχουμε φτάσει επιτέλους εδώ πέρα και η Ιωνή είναι καλή. Και εγώ καλωσορίζω όπως και ο Επίτροπος την ε, την δημοσίευση την Παρασκευή από τις ΕΠΑ του σχεδίου νέου κανόνα και ελπίζουμε να ανοίξει η αγορά βοηουκρέατος ε, των ΕΠΑ αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναφερθεί εδώ πέρα οπότε πρέπει να είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί νομίζω πως έγινε η συμφωνία αλλά πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειε και ε, από ό,τι μου λένε από τις ΕΠΑ οι κανόνες για το γαλακτικό οξύ στα σφάγια δεν τους αρέσουν πάρα πολύ, δεν είναι πρακτική και βεβαίως ε, δεν μας αρέσει αυτό να το ακούμε, αλλά έτσι μας λένε. Και άρα θα χρειαστούν κάποιες ε, διευκρινήσεις. Και επίσης ανησυχώ για το ότι χωρίς αυτές τις διευκρινήσεις δεν θα δούμε να ε, υπάρξει κινητικότητα στο ζήτημα της εξαγωγής του ευρωπαϊκού βοηού κρέατος. Οπότε ναι, επιτύχαμε πάρα πολλά, έχει σταματήσει ο εμπορικός πόλεμος, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολύ περισσότερα και από τις δύο πλευρές για να αποφεληθούμε από την κατάσταση αυτή. Τελευταία μου παρατήρηση και θα το επαναλάβω αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ακόμα. Ξέρω πως ανησυχούμε εδώ πέρα για το πόσο περίπλοκοι είναι οι κανονισμοί μας. Είναι κρίμα να μας λένε οι ΙΠΑ, γιατί μας το λένε, ε, πως είναι πολύ ε, πολύπλοκοι και δύσκολοι οι κανονισμοί μας. Οπότε θα μπορούσε ίσω να πει κάποια πράγματα ο κύριος Επίτροπος. Επίσης έχω και κάποιες ενισχύσεις για τη Ρωσία και την πρότασή τους να απαγορευτεί η εξαγωγή ζών των ζώων λόγω κάποιας αρρώστιας. Σας ευχαριστώ η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να καταναλώνουμε υπερβολικά μεγάλα ποσά όγκο ερυθρού κρέατος. Δημιουργεί κινδύνους ε, καρδιαγιακών παθήσεων και καρκίνου, λέει κάποια μελέτη. Δέχομαι παρόλα αυτά όμως το συμβιβασμό που ευρέθηκε για τη διαφορά που υπήρχε όσον αφορά ε, το βόλιο κρέα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ΕΠΑ. Σύμφωνα με τα κριτήρια τη φυτογενομικά για το βόλιο κρέα μπορεί να εισάγει ε, το κρέα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελειώνει αυτή η διαφορά επί 10 χρόνια. Και σιγά σιγά θα εισάγουν ΕΠΑ και κάποια ευρωπαϊκά ε, προϊόντα που είναι παραδοσιακά. Υπάρχει βάση δεδομένων ευρωπαϊκή για αυτά τα προϊόντα και υπάρχει και ένα προϊόν ρουμανικό, το ματζούν Λοιπόν, πώς θα εφαρμοστεί το σύστημα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα όσον αφορά τη σχέση με τη ΣΥΠΑ και πώς θα επικαιροποιηθεί το σύστημα ε, γεωγραφικών των προϊόντων που έχουν συγκεκριμένη ε, γεωγραφική προέλευση και προστατευμένα. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Για ένα λεπτό, ο κ. Λάιχτφριντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια παροιμία που λέει πως το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ε, χωρίς να ισχύει βεβαίως πάντα υπάρχουν και πράγματα που καθυστερούν και είναι στο τέλος άσχημα. Ε, υποθέτω λοιπόν πως ε, όλη αυτή η διαδικασία μετά από 15 χρόνια 15 ε, χρόνια μεγάλων συγκρούσεων με τις Ήπανα, ε, να καταλήξει με εξαγωγές και από τις δύο πλευρές οπότε είναι καλή αυτή η λύση. Τώρα έχουμε λιγότερα προβλήματα για να αποστείλουμε κάποια προϊόντα στις ΙΠΑ, τα το οποίο δεν ήταν δυνατόν πριν και θα λαμβάνουμε και εμείς ε, ποιοτικό βόλιο κρέας και θα... αν και δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον είναι αναγκαίο αυτό, αλλά βεβαίως στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει και οι δύο να υποχωρούν κάπως κάτι το οποίο συνέβη εδώ πέρα και νομίζω πως τελικά έχουμε ένα καλό ε, αποτέλεσμα. Και έχει δίκιο βεβαίω και η κυρία Μαγκίνη εδώ πέρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι θα συμβεί τελικά, αλλά νομίζω πως τελικά θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάιχτφριντ. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν κατακλείδη δεν μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι φτάσαμε σε αυτό το στάδιο. Κάποια από εσά ανέφεραν πράγματι ότι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και από τις δύο πλευρές. Για να το πούμε όμως αυτό θα πρέπει και ο πλευράς είπα να δοθεί τέρμα στο θέμα με τον σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια. Αυτό που συνέβη στις 9 Μαρτίου ήταν ένα καλό βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κυρία Μαγκίνες αναφέρθηκε στο θέμα της επεξεργασίας με το γαλακτικό οξύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ανέφερε επανειλημμένα κάθε φορά μάλιστα που είχε τη δυνατότητα να σε επαφή με τη ΣΥΠΑ έλεγε ότι αυτό το θέμα του λακτικού οξέου θα πρέπει ε, να εξεταστεί επιστημονικά και όχι σαν διαπραγματευτικό ε, στοιχείο. Όπως ζητάμε και το θέμα της ε, σπογκός να αντιμετωπιστεί επιστημονικά μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά ότι ελέγχουμε την ασθένεια και γι' αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το μέτρο σαν μη δεσμολογικό ε, ε, φραγμό. Εμεί επιλέξαμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα του γαλακτικού οξέω. Η ΕΦΣΑ έκανε μελέτε επιστημονικέ όσον αφορά την επεξεργασία ε, του κρέατος με το γαλακτικό οξύ και θα κάνει μια πρόταση επιβάσει επιστημονικής ανάλυσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι αυτό το θέμα να μην εμποδίσει τη σύναψη της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά το, τη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια, όσον αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων, οι οποίοι πρακτικά θέματα. Ίσως κάποιοι τομεί θεωρήσουν τα μέτρα δεν είναι τέλεια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τέλειο σύστημα. Αναλύουμε ακριβώς μετά από διαμαρτυρίες διαφόρων εισαγωγέων ε, να δούμε πώς μπορούμε να επιφέρουμε, περισσότερη, να ε, επιφέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και εκεί μα περιορίζει και η μέθοδος γνωστή που χρησιμοποιούμε. Η κυρία Βασέσκου που αναφέρθηκε στο θέμα της προστασίας των προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης με τις είπα ακόμα διαπραγματευόμεθα για να καταλήξουμε αμοιβαία αναγνώριση των συστήματων γεωγραφικής ένδειξης πέρα από τα εναπνευματόδη ποτά και του ίνους όπου εκεί έχουμε ειδικέ συμφωνίες αλλά Ελπίζουμε να καταλήξουμε κάπου και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ε, σε κάποια αναγνώριση αυτού του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων. Με κάποιες χώρες εξάλλου, μεγάλες χώρες όπως είναι η Κίνα, αλλά και με άλλες χώρες, στις διμερείς συμφωνίες, κάθε φορά τίθεται το θέμα αναγνωρίσεως των συστημάτων γεωγραφικών ενδείξεων και ελπίζουμε ότι το τρόπο να προχωρήσουμε και με του Αμερικανού. Ένα καλό μήνυμα ότι μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα είναι και το εξή. Πρόσφατα καταλήξαμε συμφωνία μηδέα αναγνώριση των συστημάτων μα πιστοποίηση οικολογικών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων των ευρωπαϊκών προϊόντων που μπορούν να εξαχθούν τώρα προ την αμερικανική αγορά με πιστοποίηση ε, βιολογικών προϊόντων πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώση, το ίδιο ισχύει και για τα αμερικανικά προϊόντα που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό αποδεικνύει ότι οι διαπραγματεύσει, ότι η διπλωματία στο γεωργικό τομέα, στον επιστημικό τομέα μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά στην ε, κυρία εισηγήτρια, την κυρία Κίστον Ρολ για την έκθεσή τη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που απέδειξε για μία ακόμη φορά το σύστημα συναπόφαση όχι μόνο δίνει μεγαλύτερη νομιμότητα σε αποφάσει που λαμβάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μπορούν όλα αυτά να γίνουν εγκαίρω και με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Έχει το λόγο για δύο λεπτά η κυρία Κίστοντ Ρόλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, το τελευταίο σας σχόλιο ήταν το καλύτερο. Όντως, η συναπόφαση που λειτουργεί μετά την Λισαβόνα αποδεικνύει την αξία της. Και τελικά η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο μια έκθεση για το βόλιο κρέας ε, υψηλής ποιότητας, αλλά είναι ένα μήνυμα πως οι σχέσεις μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είχαν κολλήσει λίγο, και δεν ήταν πάρα πολύ αισιόδοξε τελευταία, νομίζω μπορούν πάλι να βελτιωθούν. Και άρα είναι κάτι το θετικό συνολικά δεύτερον. Ε, κοιτώντας το μέλλον, όπως το επιβεβαιώσετε και εσείς και άλλοι, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά και βεβαίως και εδώ πέρα συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνος να προσέξουμε πολύ τις λεπτομέρειες. Πρόκειται για μία αρχή μόνο καλύτερων ε, διατλαντικών εμπορικών σχέσεων. Ένα τελευταίο σημείο, κάτι το οποίο δεν θεωρώ καθόλου αυτονόητο μετά την πολιτή μου πήρα στο Κοινοβούλιο, η εμπορική η Επιτροπή Εμπορίου και η Επιτροπή Γεωργίας κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και χαίρομαι ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Το σημείο αυτό θα το ψηφίσουμε αύριο στις 12. Ε, Περνάμε στο τελευταίο σημείο. Έκθεση επίσης της ε, κυρίας Ρόβολ για